Σα Σας ευχαριστώ. Να συγχωρείτε για την καθυστέρηση, όμως α, έπρεπε να είμαι στην Ολομέλεια. Σας ζητώ συγγνώμη που σας έκανα να περιμένετε. Έχουμε διερμηνία γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά. Είναι γλώσσες που καλύπτονται και είναι και web streamed ε, η συνεδρίασή μας. Ε, αν δεν υπάρχουν σχόλια για την ε, ημερησία διάταξη, μπορεί να εγκριθεί η ημερησία διάταξη. Τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης που έχετε στο φάκελο θα, εγκριθεί, θα εγκριθούν αύριο το πρωί στις 10, εκτός αν στείλετε παρατηρήσεις σχετικά στη γραμματεία. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, γιατί δυστυχώς η κυρία Μογκερίνη δεν μπορεί να είναι παρούσα για θεσμικούς λόγους. Πρέπει να παρακολουθεί τις ε, διαδικασίες για τη ΣΕΤΑ και ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Μιγέλη Άγχελ Μορατίνος και καθώς ο χρόνος μας πιέζει και δεν έχουμε απλή το χρόνο στη διάθεσή μας, θα του δώσω κατευθείαν το λόγο για να μας κάνει μια πρώτη εκτίμηση και να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα πρώτα μου λόγια είναι λόγια ευχαριστίας σε αυτή την Επιτροπή κοινοβουλευτική συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μια πρωτοβουλία και κάποιες ιδέες για το πώς θα δώσουμε νέα αίθηση στη δυναμική της ειρήνης, του διαλόγου και της συνεργασίας σε αυτή την πολύ σημαντική περιοχή για την Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά εδώ θα αναφέρω κάποια λόγια που έχουν να κάνουν και με τα συναισθήματά μου. Καταρχήν είμαι συγκινημένος που βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εκνέου, και ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές που είναι εδώ παρόντες και ευχαριστώ και τον Πρόεδρο. Θα ήθελα να διαβιβάσετε τα χαιρετίσματά μου στον Πρόεδρο Σούλτς και στην είπατε, πρόσωπο στην κυρία Μογκερίνη. Η βούληση και το ενδιαφέρον όλων εσάς ε, για μία περιοχή που είναι κρίσιμη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επίρου. Είμαι συγκινημένος γιατί αν δούμε τον καθρέφτη της ιστορίας και συγκεκριμένα αν δω το δικό μου παρελθόν, το δικό μου καθρέφτη που δείχνει το παρελθόν της ιστορίας και παρουσιάζω, προετοιμάζοντας αυτή την ομιλία, στη μνήμη μου είδα να περνούν διάφορες στιγμές και διάφορες πρωτοβουλίες, διάφορες προσπάθειες από τότε που με τους ε, Ιταλούς συναδέλφους ε, ξεκινήσαμε στο φόρουμ της Αλεξάνδρειας όπου οι Υπουργοί Ελενζιπέ και Μερμούσα προσπάθησαν να θέσουν σε εφαρμογή ένα πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας μέχρι την διάσημη διαδικασία της Βαρκελόνης. Φανταστείτε λοιπόν τι συνέβη τότε. Την αποκαλέσαμε διαδικασία της Βαρκελόνης γιατί κατανοούσαμε τις δυσκολίες που θα συναντούσαμε για την επίτευξη των τελικών στόχων. Συνειδητοποιούσαμε ότι η Μεσόγειος επρόκειτο να αντιμετωπίσει υπαρξιακές προκλήσεις το 1995 ήδη. Και καθώς γνωρίζαμε ότι ήταν πολύπλοκες, αβέβαιες και δύσκολες οι προκλήσεις αυτές, αντί να μιλήσουμε για ένα ειρηνευτικό σχέδιο, για ένα σχέδιο συνεργασίας, αποφασίσαμε να το ονομάσουμε μια διαδικασία, μια οδό, μια πορεία. Και κατόπιν είχαμε μια πιο φιλόδοξη διαδικασία υπό την ηγεσία της διπλωματικής πρωτοβουλίας για την Ένωση για τη Μεσόγειο και ουσιαστικά αυτό αιτιολογεί την παρουσία όλων εσάς ως ε, μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία. Και ίσως προσπάθησε να δώσει ένα ποιοτικό άλμα να κάνει ένα ποιητικό έλμα όταν οι πραγματικές συνθήκες δεν ήταν επαρκώς όριμες. Και προσπάθησε να δημιουργήσει αυτή την ένωση, να βρει αυτά τα στοιχεία ενοποίηση όταν ε, έλειπε ένα ουσιαστικό στοιχείο, μια δημοκρατία, μια εκπροσώπηση και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα διάλογο μεταξύ ίσων. Ε, για να φτάσει η γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο στη Βαρκελόνη ήταν ε, μια δύσκολη διαδικασία. Και χαίρομαι που ο φίλος μου, Φατέλ Χιλμάση, συνεχίζει από μόνος του να στηρίζει αυτή τη γραμματεία. Είναι ιδιαίτερα μόνος και ουσιαστικά κολυμπάει σε δύσκολα νερά χωρίς προσανατολισμό όμως ε, κρατά την πορεία του πλοίου. Και γι' αυτό η σημερινή συνεδρίαση μου επιτρέπει να υπονθυμίσω εν συντομία όλα αυτά τα ιστορικά βήματα για να προσπαθήσω να σας ε, ενθαρρύνω να μην αφήσετε την πολιτική βούληση να δοθεί μια νέα δυναμική ειρήνης και συνεργασία σε αυτόν τον ευρωμεσογειακό χώρο. Ο πρόεδρος τον Απρίλιο του 2003 στη Μασαλία, απευθυνόμενος στους πρόεδρους ε, των 43 κοινοβουλίων της Ευρωμεσογειακής περιοχής, στην ομιλία του είπα ότι έλειπε αυτή η πολιτική βούληση. Στην ομιλία του είπε ότι δεν ήθελε η Ένωση για τη Μεσόγειο να γίνει, σε μια, να γίνει ένας απλός Οργανισμός Ανθρωπιστικής Βοήθειας, μία ΜΚΟ, μία ένας οργανισμός σχεδίων, θα έπρεπε να υπάρχει μια πολιτική βούληση από πίσω και είχε δίκιο. Και επίσης προσέθεσε ότι ίσως αυτό που έλειπε ήταν μια ενας οργανισμος σχεδιων θα επρεπε να υπαρχει μια πολιτικη βουληση απο πισω και ειχε δικιο και επιση προσεθεσε οτι ισως αυτο που ελειπε ηταν μια στηριξη της κοινωνίας των πολιτών από αυτή την ευρωμεσογειακή κοινωνία των πολιτών που θα έκανε δικό της το σχέδιο. Με αυτά τα δύο στοιχεία ο πρόεδρος ε, Σούλτς είπε στην ε, ομιλία του το 2013, συγγνώμη το 2003, ήρθαμε σε αυτό το κοινοβούλιο και ο πρόεδρος ε, του Φόρου για τον Ευρωμεσογειακό Διάλογο μίλησε προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας και ευθύνης Όταν υπάρχει σύγχυση, όταν υπάρχει ανικανότητα, όταν υπάρχουν φόβοι, όταν υπάρχουν ερωτηματικά, τότε είναι που πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο να βρούμε λύσεις. Ο κύριος Βεναΐσα, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκο, έλεγε ότι η παγκοσμιοποίηση σκοτώνει την γειτονία. Είμαστε όλοι παγκόσμοι και δεν θυμόμαστε τους γειτονές μας. Όμως, εγώ θα έλεγα κάτι ακόμη. Αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος είναι ο χώρος όπου η παγκοσμιοποίηση συναντάται με την ε, εγκύτητα της γειτονίας και Έχουμε παγκόσμια προβλήματα, πολύ σοβαρά, όπως είναι η τρομοκρατία, η δημογραφία, η μετανάστευση, πρόσφυγες, οικονομικά προβλήματα. Εμείς, ε, οι κάτοικοι της Μεσογείου, τα ζούμε αυτά τα προβλήματα. Δεν ε, λαμβάνουν χώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι Ιταλοί, φίλοι μας, ε, τα υφίστανται, αν μιλήσουμε για τη μετανάστευση και οι επιθέσεις εμείς, κυρίως οι Ευρωπαίοι πολίτες, τις υφιστάμεθα. Και όταν πρέπει να μιλήσουμε για τη Μεσόγειο και να λάβουμε αποφάσεις για τη Μεσόγειο, φαίνεται ότι είμαστε ανίκανοι παρόλα αυτά. Φαίνεται ότι δεν έχουμε ενδιαφέρον. Εσείς που ήρθατε απόψε, ε, αυτό το θλιβερό βροχερό βράδυ του ναι, δείχνεται ενδιαφέρον. Όμως, να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αν ήταν προτεραιότητα αυτή η αίθουσα θα έπρεπε να ξεχυλίζει από κόσμο. Γιατί τα προβλήματα που θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε μας αφορούν άμεσα και μας θίγουν άμεσα ως Ευρωπαίους πολίτες. Όπως και να έχει. Αρχίσαμε ήδη να εργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια χάρη στην πρωτοβουλία ε, για, που ανέλαβε το Ίδρυμα για την πρόθεση του ευρωμεσογειακού και αραβικού διαλόγου. Και με κριτικό πνεύμα θα πω ότι για διάφορους λόγους δεν υπήρξε κριτική, έλειπε ικανότητα, βούληση, καθοδήγηση από την πλευρά των κρατών μελών, από την πλευρά των κυβερνήσεων. Όσοι ζήσαμε βαθιά τη Μεσόγειο, αποφασίσαμε να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια και προσχωρήσαμε σε μια διαφορετική πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία η οποία θέλει να αλλάξει την παραδοσιακή εστίαση που έχουμε δώσει μέχρι τώρα, που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στα προβλήματα της Μεσογείου. Δηλαδή, μια πρωτοβουλία πρέπει να είναι από κάτω προς τα πάνω και όχι το ανάποδο. Δηλαδή, οι πολίτες να αναλάβουν οι ίδιοι αυτή την αναγκαιότητα δράσης. Αν κάνουμε μια δημοσκόπηση στους ε, πολίτες ε, της ε, Μεσογείου και τους ρωτήσαμε για τη δικασία της Βαρκελόνης για την Ένωση ή τη Μεσόγειο, ούτε ένα 5% δεν θα ξέρει περί τίνος πρόκειται. Επομένως, οι πολίτες της Μεσογείου πρέπει να κινητοποιηθούν για να αναλάβουν ε, το δικό τους πεπρωμένο στα χέρια τους. Και αυτή η κοινωνία των πολιτών καθημερινά υφίσταται διάφορα δεινά και αυτό και λόγω ανάληψης δράσης από διάφορους πολιτικούς ηθήνοντες. Και είναι μια διαφορετική εστίαση, όχι βορρά-νότου. Τις πρωτοβουλίες ε, δεν πρέπει να τις αναλάβει η Ιταλική, Ισπανική, Γαλλική διπλωματία. Όχι αλλά όσοι είμαστε υπεύθυνοι και στις δύο χθες της Μεσογείου. Δεν ε, είναι ένα σχέδιο το οποίο ε, το έχουν συλλάβει στην καγκελαρία ε, ή στα πρωθυπουργικά γραφεία στο Παρίσι, αλλά πρέπει να είναι θέματα τα οποία συζητούνται από τους πολίτες και αναλύονται και στις διόχθες της Μεσογείου και να διευρυνθούν και στον αραβικό κόσμο που μας αφορά. Και να ολοκληρώσω εδώ λοιπόν. Τι έχουμε κάνει, έχουν γίνει ήδη πολλά. Ήδη υπάρχει η δομή, ήρθαμε να ενημερώσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη υπάρχει μια ομάδα ακαδημιών και ιδρυμάτων, πάνω από 50, εργάζονται για την εκπόνηση μιας λευκής βίβλου συνεργάζονται. Εγώ είχα μια ακαδημαϊκή συνεργασία που λειτουργεί και υπάρχει και μια επιστημονική συνεργασία και υπάρχει και μια πολιτική επιτροπή από πρώην Πρωθυπουργού, πρώην Υπουργών Εξωτερικών και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου και είμαστε αποφασισμένοι να κινητοποιηθούμε και να υλοποιήσουμε ένα όνειρο που έχουν όλοι οι πολίτες της Μεσογείου και ήρθαμε στο Κοινοβούλιο για να διαβιβάσουμε σε εσά αυτό το μήνυμα και έχουμε και ένα αίτημα μόνο, την υποστήριξή σας, την θεσμική και πολιτική υποστήριξή σας και την οικονομική υποστήριξη για την Επιτροπή έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη Λευκή Βίβλο. Ο τελικός μας στόχος θα είναι να ολοκληρώσουμε τη Λευκή Βίβλο, να προετοιμάσουμε τις διαπραγματεύσεις των κρατών μελών και να βρεθούμε σε ένα-δύο χρόνια σε μια θέση ώστε να είμαστε ικανοί όλοι στη Μεσόγειο και στον Ευρωπαϊκό κόσμο να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι, όπως έγινε στην πράξη του Ελσίνκη. Μια διάσκεψη που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ασφάλεια, συνεργασία, ελληνικής και ειρήνης να μπορεί να υλοποιηθεί για αυτή την ε, περιοχή του κόσμου. Αυτό είναι το μήνυμα που σας φέρνουμε από τη Γενέβη και που σας διαβιβάζω με συγκίνηση και ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Φυσικά δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με την εκκλησία σας για να υπάρχει επίδειξη αλληλεγγύης στη Μεσογείο και στον Αραβικό κόσμο. Το δικό μας ε, θεσμικό όργανο ακριβώς επί αυτών των αξώνων εργάζεται και προωθεί αυτό το διάλογο. Γι' αυτό με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αντιμετωπίζουμε τη δική σας πρωτοβουλία. Θα έλεγα να δώσουμε τώρα το λόγο στους συναδέλφους που έχουν ήδη ζητήσει. Ο κύριος Μιγελ Βιέγας, παρακαλώ καταρχήν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις για κάποια προβλήματα που αποτελούν τη συγκεκριμένη έκφανση των δυσκολιών για να καταλάβουμε σε τι βαθμό μπορεί η Λευκή Βίβλος και η Μεσογειακή Ένωση να συνεισφέρει ώστε να επιληθούν προβλήματα που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και το διάλογο ε, στον οποίο θέλουμε όλοι να καταλήξουμε. Και έχω κατά νου τη Δυτική Σαχάρα, την Παλαιστίνη. Αυτά είναι δύο προβλήματα που έχουν άμεση επίπτωση σε αυτή την περιοχή και θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω τη δική σας αξιολόγηση. Ποια είναι η κατάσταση στην Δυτική Σαχάρα, όπου υπάρχουν διάφορα επεισόδια Παραδείγματο χάρη ο αντιπρόεδρος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου που ήθελε να συμμετάσχει στην COP22 δεν του δόθηκε έγκριση γιατί είναι από την Δυτική Σαχάρα και επίσης την αποπομπή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση της κατάστασης. Και θέλω να σας ρωτήσω και για την Παλαιστίνη, όπου υπάρχουν έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνεχώς καταστρέφονται από τις βόμβες της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η συνέχιση των επικισμών, το τείχος στην Υπεριορδανία. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση για την κατάσταση αυτή και πώς θα ξεκινήσει εκ νέου ο διάλογος δεδομένων αυτών των προβλημάτων που έχουν τόσο αρνητική επίπτωση στην περιφέρεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι από μια χώρα που δεν είναι στα παράλληλα της Μεσογείου, από τη Γερμανία. Αλλά ένας πρώην πρέσβης της Γερμανίας μου ζήτησε να παρευρεθώ και να συμμετάσχω. Αν μπορείτε να επαναλάβετε γιατί δεν είχε τα ακουστικά του ο κ. Μωρατίνος. Έλεγα λοιπόν ότι είμαι από τη Γερμανία ε, και ο, ο Κέλ, πρώην πρέσβης της Γερμανίας στην την Ισία, μου ζήτησε να παρευρεθώ. Εγώ ασχολούμαι με τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχω μια ερώτηση προς εσάς. Τα σύνορα μεταξύ Ευρώπης και Βορείου Αφρικής έγιναν ε, τα πλέον θανατηφόρα σύνορα σε ολόκληρο τον κόσμο. Με απασχολεί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, των προσφύγων και το θέμα της δυνατότητάς τους να έρθουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα από τα θέματα που σας απασχολούν στη Λευκή Βίβλο. Είπατε ότι έχετε κατά νου ένα think tank, το οποίο θα καταλήξει στη Λευκή Βίβλο. Έχετε και οικονομική υποστήριξη. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το πρόγραμμα που βρίσκεται. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου προς εσάς, αγαπητέ συνάδελφε. Χαίρομαι που συνεχίζετε ε, να δουλεύετε πάνω σε αυτό το θέμα αυτού του πολύπλοκου διαλόγου Μερικέ φορέ είναι ψευδή πόθη περισσότερο παρά διάλογο, γιατί υπάρχουν και πολλές παρανοήσεις σε εμά στην Ευρώπη σχετικά με την οτροπία και την κουλτούρα και την πολυμορφία των αραβικών χωρών. Και ίσως αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους αργήσαμε να αντιδράσουμε και δεν κατανοήσαμε σωστά τα πολύ σημαντικά γεγονότα όπως την Αραβική Άνοιξη. Θέλαμε να τα ερμηνεύσουμε με το δικό μας τρόπο, αλλά τα κινήματα αυτά ήταν δικά τους. Ήταν η δική τους προσπάθεια για μια αλλαγή ζωής. Έχουμε ανταλλάξει απόψεις και στο παρελθόν. Και όλοι γνωρίζουμε ότι ακόμη και το σύντομο διάστημα της ζωής της Μεσογειακής Ενώσεως, τα προβλήματα ε, που είχαμε στις συναντήσεις μας ήταν κυρίως σχετικά με τις σχέσεις Ισραήλ-Παλαιστίνης που έθεταν και τα όρια στις δυνατότητες επικοδομητικού διαλόγου. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να μείνει ανοιχτός αυτός ο διάλογος. Δεν μπορώ να πω ότι αυτός ο διάλογος και η Μεσογειακή Ένωση έχει ήδη εκπληρώσει τις προσδοκίες μας για τις δυνατότητες ε, που πιστεύαμε ότι θα είχε. Όλοι οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάντοτε έχουν αποδώσει ύψιστη σημασία, προεδρεύουν τις συνεδριάσεις από πλευράς Κοινοβουλίου και προσπαθούν ε, να καταβάλουν προσπάθειες και για την οικονομική συνεργασία και για την ε, επιστημονική συνεργασία, συνεργασία πανεπιστημίων. Υπάρχουν δύο πανεπιστήμια, ε, ένα στη ΦΕΣ και ένα στη χώρα μου, στη Σλοβενία. Δεν φαίνεται να επαρκούν όλα αυτά. Μόλις προέκυψαν τα πραγματικά προβλήματα, ήταν προφανές ότι η Μεσογειακή Ένωση δεν μπορούσε να αποδώσει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Δεν είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει την κατάσταση. Σας ε, συγχαίρω για τις δράσεις σας. Με χαρά θα συνεργαστώ σε οποιαδήποτε ανταλλαγή απόψεων και θα προσπαθήσω και εγώ να συνεισφέρω σε κοινέ πρωτοβουλίες. Και πρέπει να πω ότι αυτό που αναφέρατε ένα είδος διάσκεψης του Ελσίνκη για τη Μεσόγειο είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, καταπληκτική ιδέα. Μια ιδέα την οποία χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Μια άλλη ιδέα που έχω αναφέρει και εγώ πολλές φορές είναι ένα σχέδιο Marshall για τη Μέση Ανατολή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση. Πρέπει τουλάχιστον να επιδιορθώσουμε τις ζημιές ε, τις οποίες βοηθήσαμε να προκληθούν στη Μέση Ανατολή και με τον πόλεμο στο Ιράκ και με άλλες καταστροφικές αποφάσεις. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι βλέπω κάποια προβλήματα ένα νέο πρόβλημα είναι τεράστιο το θέμα της ε, ρήξης της σχέσης μας με την Τουρκία και αύριο ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα θα περάσει στο Κοινοβούλιο για το τέλος των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας. Αν δεν είναι έτοιμες οι χώρες ε, να διαπραγματευθούν, τι κάνουν, αρχίζουν να πυροβολούν η μία την άλλη. Πιστεύω ότι η κατεύθυνση αυτή είναι εσφαλμένη. Όπω είπε και ο συνάδελφο προηγουμένω, το θέμα τη δυτική Σαχάρα πρέπει να συζητηθεί και πρέπει να παίξουμε εμεί κάποιο ρόλο. Ξέρω ότι είναι ευαίσθητο το θέμα των συνόρων με το Μαρόκο και καθοδόν προς τη Δυτική Σαχάρα μάλιστα με απέλασαν από το ε, Μαρόκο. Αλλά θα πρέπει ε, να αναζητήσουμε περισσότερο ενεργό τρόπο μια λύση από όλες τις πλευρές. Επίσης το πρόβλημα της Γάζας, το έχουμε ξαναναφέρει, είναι ένα ξεχασμένο πρόβλημα. Μιλάμε για ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για την πρώτη ερώτηση για, το λευκό, για τη Λευκή Βίβλο. Μια απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίλυση των πολιτικών προβλημάτων και τις εφιστάμενες σειράξεις. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη και το εσφαιλο πρόβλημα και να το συμπεριλάβουμε. Όμως, ε, από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια ικανότητα να κινηθεί η διαδικασία της Βαρκελόνης επειδή υπάρχει το Ισραηλο-Παλαιστινιακό. Όμω ε, υπάρχουν και άλλα θέματα, είτε πρόκειται για τη Δυτική Σαχαρή είτε για την Κύπρο. Ελπίζουμε να έχουμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο ενεργής διπλωματία πάντοτε ζητούσαν ενεργό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Νατώνη Κουτέρης, ο νέος Γενικός Γραμματέας, θα παίξει σημαντικό ρόλο. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι τα τελευταία έτη δεν ήταν πολύ αποτελεσματικά τέλο πάντων ήταν λιγότερο θετικά ω προ το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση κάποιων σειράξεων και κυρίως σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της Δυτική Σαχάρας. Τώρα έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχει μια νέα δυναμική, ελπίζω, μεταξύ του Μαρόκου και τη Αλγερία. Δεν είναι ακόμα πραγματική, επίσημη, όμως θα πρέπει να λάβει χώρα, να υλοποιηθεί. Και Φυσικά θα πρέπει τα Ευρωπαϊκά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι καταλήτε στην επίλυση του προβλήματο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει και πρέπει να προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε οριστικά. Συμφωνώ μαζί σα λοιπόν. Θα πρέπει να αναλάβουμε δεσμεύσει, θα πρέπει να εμπλακούμε και θα πρέπει να δώσουμε στον Γενικό Γραμματέα τη δυνατότητα να σημειώσει πρόοδο στο πρόβλημα τώρα για την Παλαιστίνη και θα επανέλθω από τις διαδικασίες. δυστυχώς είναι μια ξεχασμένη σύραξη. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζετε ότι στις 29 Οκτωβρίου είχαμε την επέτειο των 25 χρόνων από την ιστορική διάσκεψη, την ειρηνευτική διάσκεψη στη Μαδρίτη. Ακούσατε κάποια αναφορά, ακόμη και στη χώρα μου, Κάποια δραστηριότητα, κάποια εκδήλωση. Παρ' όλα αυτά, στο διεθνή τύπο ούτε μία λέξη δεν γράφτηκε. Πρόκειται για μία εγκαταλελειμμένη ειρήνη και μία ξεχασμένη ιστορική στιγμή. Δεν είναι δυνατόν. Δεν θα εξαφανιστεί το πρόβλημα. Η Παλαιστίνη δεν θα εξαφανιστεί. Είναι εκεί. Και εμείς, οι Ευρωπαίοι, θα έχουμε μέγιστη ευθύνη γιατί δεν γνωρίζουμε τι δράση θα αναλάβει και τι αποφάσεις θα λάβει η Αμερικανική κυβέρνηση και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι θα περιμένει να επιληθεί ως διαμαγεία στο πρόβλημα. Δεν έχουμε συμφέροντα συζητούσα με έναν ε, παιδικό μου φίλο, τον κύριο Ιβολέρ, και λέγαμε ότι το Παλαιστινιακό πρόβλημα αποτελεί την ε, κύρια αιτία των προβλημάτων στη Μέση Ανατολή. Αν δεν υπάρξει ειρήνη μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ θα έχουμε άλλες αισθήσεις κρίσης και αστάθειας. Τι πρέπει να περιμένουμε για την ε, λύση των δύο κρατών στα πλαίσια της δικής μας πρωτοβουλίας και στα δικά μας έγγραφα. Το Ισραηλο-Πανεπιστημιακό πρόβλημα είναι ύψιστη προτεραιότητα. Όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Διπλωματία θα πρέπει να προετοιμαστούν. Εδώ, στις 5 Νοεμβρίου το είδατε αυτό το θέμα και θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις, λέμε στα ισπανικά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εμπλακεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, για τη Γερμανίδα βουλευτή. Σας ευχαριστώ για το σχολείο σας. Φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μέρος της Λευκής Βίβλου. Ήδη η δουλειά που έγινε από την ακαδημαϊκή μας ομάδα, από αυτά τα 43 think tank, συμπεριλαμβάνουν ε, ως προτεραιότητα, συμπεριλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως προτεραιότητα. Αυτό είναι μια κοινοτομία γιατί οι ε, άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και αυτό είναι το νόημα των λαών και των κοινωνιών. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αναπτύξουμε αυτή την ικανότητα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι ένας από τους πυλώνες της πρωτοβουλίας ε, σε όλες τις καταστάσεις, ανά πάσα συνθήκη. Το ίδιο και με το προσφυγικό. Τι μπορούμε να πούμε τώρα στην Ευρώπη για τους πρόσφυγες. Ακόμη και ο όρος πρόσφυγας είναι ένα αμάγαλμα. Μπερδεύουμε τους όρους οικονομικός μετανάστης, πρόσφυγας. Ένας πρόσφυγας πρέπει να προστατεύεται, να χέρι προστασίας. Γιατί διαφεύγει από το χάος, από το διωγμό και η ζωή του απειλείται. Εμεί οι Ευρωπαίοι θα χάσουμε τις αξίες μας. Φυσικά και όχι. Θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που θα υπερασπίσουμε και θα αντιμετωπίσουμε νομικά αλλά και ηθικά την προσφυγική κρίση. Τώρα, για όσα είπα ο Ήβο. Ναι, υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν καταλάβαμε τι σήμαινε η Αραβική Άνοιξη. Στην αρχή είχαμε μια θετική ανταπόκριση, στη συνέχεια υπήρχε ένα μπέρδεμα. Γιατί? Γιατί προσπαθήσαμε να αναλύσουμε μια κατάσταση χωρίς να υπάρχει προοπτική. Εσύ είσαι Σλοβαίνος, εγώ είμαι Ισπανός, δεν ήμασταν στην την Ισία, στην Αίγυπτο. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε, διαβάζουμε, καταλαβαίνουμε κάποια στοιχεία, αλλά δεν είμαστε εκεί, ούτε είμαστε οι άνθρωποι αυτοί. Είναι διαφορετικά τα προβλήματα. Η νέα προσέγγιση που θέλουμε να έχουμε είναι να γίνεται από κοινού η ανάλυση προκειμένου να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις. Αν ε, σου εξηγήσει κάποιος γιατί τώρα πρέπει να γίνουν εκλογές ή γιατί πρέπει να καθυστερήσουν οι εκλογές, γιατί δεν είμαι έτοιμος και αν υπάρξουν εκλογές θα υπάρχει νίκη Ισλαμικού κινήματος και τα λοιπά, δεν είναι πολύ καλύτερη από εμά. Αλλά εμείς λέμε όχι, εκλογές αύριο. Υπό ποιες συνθήκες θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Με ποιες εγγύσεις. Ποια είναι τα πραγματικά κριτήρια για να έχουμε επιτυχή εκλογική διαδικασία. Όχι, εμείς όμως στην Ευρώπη λέμε αμέσως θέλουμε εκλογέ και μετά το αποτέλεσμα δεν μα ικανοποιεί. Έτσι λοιπόν ε, λέμε όχι, δεν δεχόμαστε το εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να συζητούμε μαζί τους, να τους βοηθάμε. προκειμένου να προωθούν τις δικές τους ε, ικανότητες, προκειμένου να προχωρήσουν μπροστά. Και αυτό λοιπόν είναι μέρος της Λευκής Βίβλου. Τώρα και πάλι για το την ε, Παλαιστίνη. Ευχαριστώ που με ενημέρωσες ε, για την ε, πρωτοβουλία να έρθουν νέοι άνθρωποι από τη Γάζα στο Κοινοβούλιο. Να το κάνετε αυτό. Πρέπει να τους δώσουμε ουσιαστικά μια ελπίδα, να τους υποστηρίξουμε να τους δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε, πρέπει να τους δείξουμε ότι η Ευρώπη δεν τους εγκαταλείπει. Σας ενθαρρύνουμε λοιπόν να ακολουθήσετε αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά ναι, η Ένωση για τη Μεσόγειο, συμφωνώ με την άποψή σας ε, ότι δεν είναι εδώ το θέμα του ρόλου του Γενικού Γραμματέα είναι το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει πολιτική υποστήριξη. Κανείς ε, δεν ε, υποστηρίζει ε, τον Παλαιστινό Πρόεδρο. Ναι. Ποιος του δίνει κάποια καθοδήγηση. Δεν θέλουμε τώρα μια πρωτοβουλία για να αντικαταστήσουμε την Ένωση στη Μεσόγειο. Όχι, απλώς θέλουμε να την ενισχύσουμε, να την προσαρμόσουμε στου νέου καιρού, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα project. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητές μα. Αναφερθήκατε στο σχέδιο Μάρσαλ για την οικονομική στήριξη στη Μεσόγειο. Βεβαίως, συζητάμε την ανάγκη ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού για την Μεσόγειο. Δημιουργήσαμε ένα τέτοιο μηχανισμό για την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά όταν ε, μιλήσαμε με τον Υπουργό Οικονομικών να δημιουργηθεί ένα παρόμοιο εργαλείο για τη Μεσόγειο, είπαν όχι, αν το είχαμε δημιουργήσει αυτό πριν 10 χρόνια. Και τότε δεν είχαμε κάνει του υπολογισμού, αλλά ίσω τώρα θα το κάνουμε στη Λευκή Βίβλο. Πόσα δαπανώνται τώρα σε μέτρα ασφαλείας ε, για να γίνονται περιπολίες στη θάλασσα για να προστατεύουμε τους εαυτούς μας. Αναφέρατε το παράδειγμα το πόσα πρέπει να δαπανούμε. Και αντιθέτως ε, θα έπρεπε να βοηθούμε τις ε, μικρές και μεσές επιχειρήσεις να δημιουργούν θέσεις εργασίας, όμως ε, είπαν όχι οι Υπουργοί Οικονομικών. Και συνεχίσαμε και τίποτα δεν έγινε. Και μετά εκπλησόμαστε όταν έρχονται οι πρόσφυγες ε, στη Βιέννη και στο Βερολίνο όταν έρχονται στην Ιταλία. κανένα δεν τον ενδιαφέρε όταν πήγαιναν στην Ιταλία. Πρόσφυγες μόνο την Ιταλία αφορούσε. Ενώ όταν έφτασαν στο Βερολίνο μα αφορά όλου το θέμα. βεβαίω και πολύ καλά. Καλωσορίσατε στο να ενδιαφέρεστε όλοι. Όμως πρέπει να κινηθούμε και να λάβουμε τι σωστέ αποφάσεις. Και κάτι για την Τουρκία. Συμφωνώ μαζί σα απόλυτα. Δεν ε, συμφωνούμε για το συμβαίνει με το τι συμβαίνει στην Τουρκία βεβαίω. Όμως τώρα παραποτέ χρειάζεται ανάληψη ευθύνη, συμμετοχή, όχι πάγωμα, όχι αναστολή. Αυτό που χρειάζεται η Τουρκία είναι διάλογο και συμμετοχή και κατόπιν θα δούμε τι θα πρέπει να γίνει ή όχι. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις, αλλά η δική μου προσωπική απόψη είναι ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά εμπλοκή από τη δική μας πλευρά και κατόπιν θα λάβετε τις αποφάσεις, δεν τους δώσετε πράσινη κάρτα. Αλλά αυτή είναι η δική μου προσωπική εμπειρία στην διπλωματία. Σας ευχαριστώ ότι πρέπει να εμπλακείτε. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Μωρατίνος. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Όμως ε, θα έλεγα να συμμετέχει στη συζήτηση και πριν Κουλέκη που είναι ο πρόεδρος ε, του Ιδρύματος και θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω τι ακριβώς περιμένει το Σύνδρυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποιες μπορεί να είναι οι κοινέ μας προτεραιότητες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. το Ίδρυμα για την Πρόθεση του Μεσογειακού και Ευρωαραβικού Διαλόγου θέλει να προσεγγίσει το μεσογειακό και ευρωαραβικό ζήτημα με διαφορετικό τρόπο. Έλεγα λοιπόν ότι το Ίδρυμα για την Προώθηση του Μεσογειακού και Ευρωαραβικού Διαλόγου δημιουργήθηκε για να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια απάντηση σε ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και χρόνια χωρίς να έχει βρεθεί λύση. Έχουμε καταγράψει τρεις αποτυχημένες προσπάθειες το 1994, το 1995, το 2008 παρά την καλή θέληση που είχαν δείξει οι κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων εκείνων. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να εξετάσουμε το τι έγινε στις διαπραγματεύσεις αυτές και να προσπαθήσουμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνας, διαπιστώσαμε ότι στις διαπραγματεύσει αυτές και ιδίως στη διαδικασία της Βαρκελώνας δεν είχαμε ακούσει προσεκτικά εκ των προτέρων την κοινωνία των πολιτών. Θελήσαμε να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα χωρίς να ζητήσουμε τη γνώμη των ενδιαφερομένων πληθυσμών. Σήμερα και αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε αυτό το Ίδρυμα, πιστεύω ότι δεν μπορούμε πια να λαμβάνουμε τέτοιες αποφάσεις χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών. Διαπραγματεύσεις ε, που προσπαθούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη συνεργασία που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει οπωσδήποτε να περνούν από ένα στάδιο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών. Και από αυτή τη βάση μπορούν οι κυβερνήσει στη συνέχεια να υποβάλουν προτάσει. Μέχρι τώρα αυτό δεν είχε γίνει. Και σήμερα, στον Μεσογειακό Ευρωαραβικό Διάλογο, έχουμε την εντύπωση ότι φοβόμαστε την αποτυχία και γι' αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Και αυτή η αδράνεια είναι πραγματικά τρομερή σήμερα μια στιγμή που τη χρειαζόμαστε όσο ποτέ. Χρειαζόμαστε προτάσεις για να δείξουμε ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικέ λύσεις έναντι των κινήματα που είναι επικίνδυνα για τη δημοκρατία μας. Είναι λοιπόν επίγον το να αναλάβουμε δράση και πιστεύουμε ότι μιας και σε μια δύσκολη στιγμή ε, ε, ξεκινήσαμε με τη διάσκεψη του Ρίο η διάσκεψη του Ρίου δεν θα είχε ποτέ γίνει κατά αυτόν τον τρόπο αν ε, υπήρχε μια λευκή βίβλος που θα επέτρεπε στις κυβερνήσεις ε, να διαχειρίζονται τα προβλήματα που προέκυπταν. Αυτό που έγινε είναι ότι δημιουργήθηκε μια επιτροπή ε, που οργάνωσε μία ακρόαση σε παγκόσμιο επίπεδο για να καταγράψει τα βασικά προβλήματα για το περιβάλλον. Οι περισσότερες κυβερνήσεις εκείνη την εποχή δεν θεωρούσαν το περιβάλλον ως κάτι το ανησυχητικό και από αυτή την λευκή βίβλο προέκυψαν γύρω στις 20 προτάσεις και μία πρόταση ήταν να συγκληθεί αυτή η παγκόσμια διάσκεψη για το περιβάλλον που έγινε το 1992. Χωρίς αυτή τη λευκή βίβλο δεν θα γινόταν καν συζήτηση για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή σήμερα. Η αλλαγή του κλίματος ήταν μία από τις προτάσεις που προέκυψαν το αναφέρω για να σας εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι να αναλάβουμε κάποια δράση. Και μάλιστα διότι από το 2011 η Ευρώπη δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα των νέων που ξεσηκώνονταν. Πάρα πολλές διεκδικήσεις που δεν έτυχαν καμιάς απάντησης. το οποίο προτείνουμε είναι μια διαδικασία βήμα-βήμα να συντάξουμε μια λευκή βίβλο που θα καταγράψει όλες τις ανησυχίες του αραβικού και ευρωαραβικού κόσμου και με βάση τις προτάσεις αυτές θα ζητήσουμε στη συνέχεια από τις κυβερνήσεις να λάβουν θέση και να ξεκινήσουν πλέον μια πολιτική διαπραγμάτευση γύρω από αυτές τις προτάσεις, ξέροντας ότι αυτές οι προτάσεις υποστηρίζονται από τους εν λόγω πληθυσμούς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα είδος πράξης του Ελσίνκη, όπως ανέφερε ένας ευρωβουλευτής προηγουμένως, που θα μπορούσε να είναι η πράξη της Τίνιδας ή η πράξη μιας αραβικής, άλλης αραβικής πόλης. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο κάτι τέτοιο αυτή η λευκή δίβλος πώς θα γίνει. Όπως είπε ο πρόεδρος Μορατίνος, υπάρχουν γύρω στις 40 ευρωαραβικές ε, ενώσεις που θα θέλουν να συμμετάσχουν και ξέρουμε και άλλα 20 πανεπιστημιακά Ινστιτούτα που θα θέλουν να συμμετάσχουν. Θα είναι πολύ περισσότεροι δηλαδή οι συμμετέχοντες φορείς και στο πεδίο αριστείας του ο καθένας μπορεί να προτείνει κάτι κατόπιν διαβουλεύσεων με την κοινωνία των πολιτών. Η Λευκή Βίβλος θα έχει ένα κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα θέλουν να συμμετάσχουν. Θα υπάρχει και ένα κεφάλαιο για το νερό και ένα κεφάλαιο για την ενέργεια, ένα κεφάλαιο για τις μεταφορές, για το περιβάλλον, για τις γυναίκες, για τη δημοκρατική διαδικασία, για την ασφάλεια πολλά κεφάλαια που όλα μαζί θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας στη συνέχεια θα μπορούν οι κυβερνήσεις να διαπραγματευτούν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θα δημιουργήσουμε κάποια καινούργια δομή. Προτείνουμε τρόπους διαπραγμάτευσης και αυτές οι μέθοδοι διαπραγμάτευσης ήδη υπάρχουν αλλά θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πρόοδο. Έχει βέβαια κάποιο κόστος η Λευκή Βίβλος, το οποίο είναι ελάχιστο αν σκεφτούμε όλες τις υπόλοιπες δαπάνες. Θα χρειαστούν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ και με αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε δύο χρόνια, το 2017-2018, αυτό υπολογίζουμε μαζί με, όλα, με όλους τους πανεπιστημιακούς φορείς που ήδη ασχολούνται με τη Λευκή Βίβλο, θα μπορούμε να θέσουμε επιτάπητος κάποιες προτάσεις που θα μπορούν οι διαπραγματευτές να τη συζητήσουν στη συνέχεια. Δεν δημιουργούμε λοιπόν, τονίζω, καμία καινούρια δομή. Μέχρι τώρα, απαντώντας σε μια ερώτηση, δεν έχουμε κάνει επισήμως ε, αίτηση ε, επιδότησης. Έχουμε ένα μνημόνιο για να διαπραγματευτούμε με τις αρμόδιες αρχές που θέλουν να υποστηρίξουν την προσπάθειά μας και είμαστε στη διάθεσή σας εάν επιθυμείτε να βοηθήσετε. Στην Γενέβη έχουμε μια γραμματεία που θα πρέπει βέβαια να αναπτυχθεί για να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα αιτήματα. Υπάρχει ήδη ένα πανεπιστήμιο που θέλει να αναλάβει να συντονίσει τα 60 περίπου πανεπιστήμια που θα συμμετάσχουν στη Λευκή Βίβλο. Αυτό το οποίο προς το παρόν δεν έχουμε είναι η πολιτική βούληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρεσβευτά. Μικρόφωνο παρακαλούμε για τον Πρόεδρο. Τρία άτομα έχουν ζητήσει ακόμη το λόγο. Θα έλεγα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ροντρίγκε καταρχή. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έτσι λοιπόν να αυτορυθμιστούμε. Ευχαριστώ. Δεν θα προσπαθήσω να μιλήσω ισπανικά. και είναι καλό να ακούμε ότι αυτό που μας είπες δεν φαίνονται τόσο επίσημα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα λόγια αυτά. Μου δίνουν δύναμη και ελπίδα και είναι σημαντικό. Όπως ε, είπε η Μεσόγειος είναι πρόβλημα όλων μας. Όταν μιλάμε για τη Μεσόγειο πηγαίνουν πολύ αργά τα πράγματα. Έχουμε το πρόβλημα της δημαγωγίας, του λαϊκισμού. Δεν θα σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί οι συνάδελφοι το έκαναν ήδη. Ανησυχώ για την κατάσταση στην Τουρκία πάρα πολύ. Μια άλλη ερώτηση που είχα, είχε να κάνει με τη Λευκή Βίβλο, δεν θα το αναφέρω. Απλώς θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με κάτι που είπατε. Είπατε ότι οι πρωτοβουλίες για διάλογο θα πρέπει να γίνονται από κάτω προς τα πάνω από τους πολίτες και ότι αυτοί θα πρέπει να γράφουν την ιστορία τους. Όμως είναι τόσο δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί προσπαθούμε να το κάνουμε σε κάποιες περιοχές. Εγώ προέρχομαι από μια μικρή περιφέρεια, τη Μαδέιρα, στην Πορτογαλία, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούμε τον αραβικό κόσμο στις χώρες μας. Έτσι λοιπόν, ποια συμβουλή μπορείτε να μας δώσετε και ποια σχέδια θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε με τους πολίτες γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, να συμμετέχουν οι πολίτες στο διάλογο αυτό. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο παρακαλούμε για τον Πρόεδρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ τέλεια να σας έχουμε εδώ. Αμφιβάλλω αν υπάρχει κάποιος στην Ευρώπη που να γνωρίζει καλύτερα την κατάσταση στη Μεσόγειο και πραγματικά και εγώ λυπάμαι που δεν είναι πιο γεμάτη η αίθουσα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Θα κάνω τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη πάνω κάτω το σχολείο σας, αλλά θα ήθελα κάποια ανδάθυνση. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να ξαναλειτουργήσει η γραμματεία της ε, Ένωσης για τη Μεσόγειο, είναι στη Βαρκελόνη, όπως ε, είπες ε, και εσύ είναι εξαιρετικός πρεσβευτής, εξαιρετικός γραμματέας, ο αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει και νομίζω ότι είναι ο μόνος τόπος όπου κάθονται στο ίδιο τραπέζι το Ισραήλ και η Παλαιστίνη. Και αυτό είναι ήδη κάτι πολύ σημαντικό. Όμως τι μπορούμε να κάνουμε για να ξαναλειτουργήσει. δεύτερη ερώτηση για την Αραβική Άνοιξη. Θα αναφέρω μια μικρή ιστορία πριν τρία χρόνια. Όταν ε, δεν ήμουν πρόεδρος, ε, έδωσα μια συντευξή ε, μαζί με τον σημερινό πρόεδρο της και του είπα κύριε πρόεδρε, η Αραβική Άνοιξη μου πήρε το χέρι και μου είπε κύριε βουλευτή μη λέτε η Αραβική Άνοιξη αλλά να πείτε ο Αραβικός χειμώνας. Επομένως, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που υπάρχει. Και πώς βλέπετε αυτή την δημοκρατική ανάπτυξη ε, των χωρών αυτών. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να επιβάλλουμε τους δικούς μας ρυθμούς, αλλά αυτές οι χώρες θα πρέπει να διαλέξουν το δικό τους ρυθμό, που είναι πιο κατάλληλος για αυτές. Και κάποια τελευταία ερώτηση, που είναι δύσκολο όσο το ξέρουμε, τι θα γίνει με την Προεδρία Τραμπ. Αυτό μπορεί να αλλάξει εντελώς την εξωτερική πολιτική. Και πώς πιστεύεις ότι θα επηρεάσει η θητεία του Τραμπ στην μεσογειακή πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παρνιό για την τελευταία παρέμβαση. Πολύ σύντομα, γιατί περνάει η ώρα και ήδη έχετε απαντήσει σε αρκετές ερωτήσεις συναδέλφων. Εξάλλου συναντηθήκαμε και πριν από τη συνεδρίαση και ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις. Βλέπουμε ότι η βάση στα προβλήματα που έχουμε είναι να δημιουργηθεί ένας νέος διάλογος όπως αυτόν, αυτός που περιγράφεται στη Λευκή Βίβλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής της Ένωσης για τη, για τη Μεσόγειο μια λαμπρή ιδέα γιατί συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το διάλογο 43 χώρες συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, της Παλαιστίνης αλλά και της Τουρκίας που όπως είπαμε μας ενδιαφέρει για την ε, επίκαιρο το θέμα της συζήτησης που θα γίνει στο Κοινοβούλιο. Αυτό που λείπει είναι ο πολιτικός διάλογος, όπως είπε ο Πρέδης και δυστυχώς από το 2008 δεν υπάρχει πολιτική βούληση από πολλά κράτη-μέλη της Μεσογειακής Ένωσης που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη. Μέσα στην παγκόσμια έλλειψη τάξης και βλέποντας ε, τον ανερχόμενο εθνικισμό και βλέποντας ε, και την άνοδο του Ισλάμ, οι προτάσεις σας βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση για προβλήματα όπως η μετανάστευση, η τρομοκρατία, η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, ο εξηλεκτρισμός της Αφρικής, ε, το πρόβλημα της ίδρευσης. η αυριανοί πόλεμοι θα είναι πόλεμοι που έχουν σχέση με το νερό, που σιγά σιγά αρχίζει να σπανίζει. Όλα αυτά είναι ζητήματα για τη Μεσόγειο. Τι να κάνουμε λοιπόν. Η ευρωπαϊκή διπλωματία ε, μέσω της κυρίας Μογκερίνη έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Δημιουργήσατε λοιπόν μια πολιτική επιτροπή. Αυτή τη βούλησή σας μας ανακοινώνεται. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορούμε να πιέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτω ώστε αυτή η πολιτική επιτροπή την οποία εσείς θέλετε να δημιουργήσετε να έχει μια πολιτική δύναμη όχι μόνο για τις προτάσεις ε, των δράσεων που αναλαμβάνετε αλλά επειδή πολύ σωστά είπατε κύριε Υπουργέ από γεωπολιτικής άποψης η επίλυση ε, της ε, συγκρουση ισραηλ Ισραήλ-Παλαιστίνη βρίσκεται στην καρδιά όλων των προβλημάτων. Πώ μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και για μια ειρηνευτική προσπάθεια Ισραήλ-Παλαιστίνη. Με τον άλλον Μπενμέρ, καθαναθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νέα Υόρκη και με τον Πιάχ Βημό από την πλευρά τη Γαλλική Διπλωματία αναλάβαμε κάποιε πρωτοβουλίε όπου όμως δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα με την πρωτοβουλία σας και με την πείρα σας όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε έναν εξέχοντα ρόλο με συγκεκριμένες προτάσεις που θα μας ανακοινώσετε εσείς. Ε, Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη γιατί καθυστέρησα να φτάσω και δεν άκουσα όλα όσα υπόθηκαν. Όμως ε, θα να κινδυνεύσω να κάνω κάποιο λάθος ε, και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για το ρόλο της Γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο, για τον πολιτικό ε, ουσιαστικά ρόλο που έχει. Δηλαδή, πέρα από ότι προωθεί και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα σχέδια, νομίζω ότι υπάρχει και ένα πραγματικό έλλειμμα πολιτικού χαρακτήρα για έναν οργανισμό που πιστεύουμε ότι έχει σχεδιαστεί γι' αυτό καταρχήν. Η δεύτερη ερώτηση, αν το έχετε ήδη πει, δεν χρειάζεται να ξαναπαντήσετε για την Τουρκία. Και μάλιστα χτες σε αυτό το κοινοβουλίο είχαμε την ιωστή συζήτηση για την Τουρκία και προσθέσαμε ουσιαστικά και μία πιο ε, επιθετική θέση, αν θέλετε, για το ποια θα είναι η θέση η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι είμαστε εν ώψη μιας ε, προοπτικής πραγματικής ρήξης. Έχει ουσιαστικά λήξει το ζήτημα αυτή η ψευδέστηση και σε τι κάναμε λάθος, γιατί νομίζω ότι και εμείς κάναμε λάθος και δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι η ευθύνη η δική μας αιτιολογή και αυτά που βλέπουμε σήμερα στην Τουρκία και κάτι ακόμη σε σχέση με τη σημερινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται ότι είναι ουσιαστικά η Ευρώπη αυτομπλοκάρεται στο θέμα της ε, άμυνας και της ασφάλειας Όμω, θα έπρεπε να επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό, δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε και στην πολιτική Ευρώπη, η οποία θα πρέπει με τη δική της ε, επιρροή ε, ουσιαστικά να επηρεάζει τα δρόμενα σε αυτή την περιοχή και με την ηγετική της θέση. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον Πρόεδρο Ρατίνος, υπενθυμίζοντα ότι πολλέ από τι παρατηρήσει που έγιναν από του συναδέλφου. εντάσσονται στο πνεύμα που θα πρέπει να διακατέχει τη συνέλευση για τη Μεσόγειο. Εμείς βρισκόμαστε τώρα σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί πολλές χώρες ε, έχουν, ε, σε πολλές χώρες έχει αλλάξει και η πολιτική σκηνή στην άλλη της Μεσογείου. Και φυσικά αυτό μας βάζει όλους μας σε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ταυτόχρονα Προσπαθούμε ουσιαστικά να κρατάμε ζωντανή την ελπίδα στην Ευρώπη και πώς θα τροποθετήσουμε αυτή την ελπίδα αν δεν έχουμε ε, σχέση με την κοινωνία των πολιτών, με τις ενώσεις, με τμήματα της διπλωματίας που να μπορούν να μας βοηθήσουν. Φυσικά όλα αυτά για μας είναι μόνο η επαρχή ενός διαλόγου και φυσικά θα συνεχίσουμε το διάλογο αυτό και κυρίως ε, θα λάβουμε και δικά σας ζητήματα για να σας βοηθήσουμε στο έργο σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία Ροντρίγιας. Η Τουρκία. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να απαντήσω και στον κύριο Μαραγάλη. Η σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κάτι καινούριο, είναι πάρα πολύ παλιά η σχέση. Ήταν υποψήφια χώρα, δεκαετία του 60 και ακόμα εδώ είναι. Φυσικά. Τώρα έχουμε μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση με τον πρόεδρο Ερντογάν και τη στάση του και τις δράσεις του. Πολλά ερωτηματικά. για τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Κατανοώ ότι θα πρέπει να συζητηθούν αυτά και να είναι ουσιαστικά μέρος μιας αναλυτικής συζήτησης εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι απαραίτητο αυτό. Όμως, η δική μου εμπειρία για τη σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι έχουμε κάνει πολλά λάθη την τελευταία δεκαετία. Τότε ε, οι Υπουργοί Εξωτερικών ανήκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω αν η σημερινή εξέλιξη είναι καλύτερη ή χειρότερη, απλώς ήταν ένα σχόλιο. τότε συλλογικά πήραμε τη στρατηγική απόφαση να προσελκύσουμε την Τουρκία προς την Ευρώπη και κάποιες χώρες τότε αποφάσισαν να παγώσουν τις διαπραγματεύσεις. Θυμάμαι ότι το τελευταίο κεφάλαιο που άνοιξε πριν από την προσφυγική κρίση άνοιξε υπό, υπό την Ισπανική Προεδρία το 2010 άνοιξαν εκεί δύο τελικά κεφάλαια με την Τουρκία. Από το 2010 μέχρι το 2015 τίποτα. Και μετά έρχονται οι πρόσφυγες και πρέπει να λύσουμε το προσφυγικό ζήτημα. Και τώρα ναι. Ερντογάν, φίλε μου, Αχμέντα Βούντογλου, έλα να διαπραγματευτείς με την καγιλάριο Μέρκελ. Και μετά οι Τούρκοι βρίσκονται σε ισχυρή θέση και λένε να αυτά χρειάζομαι εγώ για τη συμφωνία. Και οι Ευρωπαίοι τελικά συμφωνούν. Γιατί τα επενθυμίζω τώρα όλα αυτά. Γιατί αύριο μεθαύριο πρέπει να αποφασίσουμε να παγώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Σήμερα όμως συνομιλούμε με την Τουρκία, αλλά ίσως σε τρεις μήνες θα χρειαστούμε την Τουρκία και το τίμημα της Τουρκίας θα είναι υψηλότερο και θα γονατίσει η Ευρώπη. Σουλτάνε, σε παρακαλώ να συμφωνήσεις ε, με τα επιχείρηματα. Αντίθετα όμως, αν διαπραγματεύεσαι, αν είσαι τέρος, αν θες να κερδίσεις όχι μόνο τον Ντογκάν, αλλά και την ε, κοινωνία των πολιτών, γιατί η κοινωνία της Τουρκίας θέλει να είναι ευρωπαϊκή, θέλει να έχει αξίες. Φυσικά θα πρέπει να σκηθεί και κάποια κριτική, όμως το καλύτερο είναι να παγώσει διαδικασία και να επιπλακούμε από την όλη διαδικασία, όχι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συμμετέχει σε μια διαδικασία, να είσαι σκληρός, όμως θα πρέπει να διατηρήσεις μια διαδικασία. Εκεί είναι ο Μοχλός. Εσύ πρέπει να είσαι αυτός που κινεί τα νήματα προκειμένου να αλλάξει η Τουρκία, προκειμένου να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπενχάγης και να τηρήσει τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Αυτά έχω να πω για την Τουρκία. Κύριε Ροντρίγε, αναφερθήκατε στην κοινωνία των πολιτών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και <laughs> είπα αναφερθήκατε και στη Μαδέρα. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αλλά δοκιμάζουμε ένα νέο τρόπο. Αυτό με το think tank. Φυσικά προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτό το διάλογο μέσω του δυνατόν περισσότερους ανθρώπους Προσπαθούμε να απευθυνθούμε σε όσο το δυνατό περισσότερους και να έχουμε ουσιαστικά και ένα πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι δύσκολο δεν θα προσπαθήσουμε. Αν αποτύχει μια φορά, πρέπει να επιμείνει Και δεύτερη φορά. Και αν επιμείνει και δεύτερη φορά, πρέπει και τρίτη φορά. Και πρέπει να βρει νέου τρόπου. και οδού. Έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. για το φίλο μου και συμπατριώτη μου, τον Σαντιάγο, με τον οποίο συνεργάστηκα πολύ στενό όταν ήμουν υπουργό στην Ισπανία. Να του πω ότι τον ευχαριστώ για τα λόγια του. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και πώς ε, θα ενισχύσουμε τη γραμματεία της από εδώ και στον κύριο Μαραγάλ ταυτόχρονα. Πώς θα τη δώσουμε μια πολιτική αποστολή. Εγώ έχω διάφορε ιδέε. και νομίζω ότι με την νέα κυβέρνηση που τώρα είναι κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα θα πρέπει η δική μας χώρα να αναλάβει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά εγώ νομίζω ότι και με την πρωτοβουλία που παρουσιάσαμε εδώ. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ο κοινό μας φίλος, ο Φατάλης Ιχμαπ, ε, θα καλούσε μια συνεδρίαση των χωρών που θεωρούν ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει νόημα. Και να είναι αυτοί, αυτοί που θα μπορούσαν να προωθήσουν ένα διάλογο και να κληθεί μια συνεδρίαση υπουργών των χωρών που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, ότι κάτι πρέπει να κάνουν για τη Μεσόγειο και να μην είναι μια συνεδρίαση δίωρη, όπως αυτή που έλαβε χώρα για να γιορτάσουμε την 20η επέτειο της Βαρκελόνης, της δημιουργίας της διαδικασίας Βαρκελόνης και της Γραμματείας. Όχι. Εγώ ξέρω ότι είναι πολύ απασχολημένοι οι υπουργοί. Όμως, έχει χαθεί το νόημα της πραγματικής διπλωματίας. Χρειάζεται χρόνος, ώρες, συζήτηση, προτεραιότητες. Δεν θα ζητήσω τώρα να κάνουμε μια παρόμοια συνάντηση όπως έγινε το 1919 και είχαμε τους προέδρους να διαπραγματεύονται για 7 μήνες. Όχι, δεν ζητώ κάτι τέτοιο, αλλά σα ζητώ μια μισή μέρα να μείνουν και να διαπραγματευτούν με τους συνομιλητέ τους. Μια μισή μέρα, αν είναι προτεραιότητα στην ατζέντα των Υπουργών. Δεν τους λέω να δουν τι γίνεται στην Καραϊβική, αλλά τι συμβαίνει στα μέσα σύνορά τους, στη Μεσόγειο. 24-48 ώρες, μόνο αυτό. Και η γραμματεία θα έπρεπε να ξαναλάβει, αναλάβει ηγετική θέση γιατί αυτοί οι υπουργοί θα έδιναν στη γραμματεία αρμοδιότητες, εξουσίες, μεγαλύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά θα πρέπει να έχει και πολιτικό πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι απλώς να διαχειρίζεται κάποια έργα. Η Ένωση για τη Μεσόγειο είχε δύο νέους πυλώνες όταν ε, δημιουργήθηκε και την πρότεινε ο πρόεδρος Σαρκοζή. Το ένα ήταν οι συνοδικορφείς, Πολιτικές. Κάθε δύο χρόνια σχεδιαζόταν ότι θα υπήρχε μια τέτοια συνοδικορφής και ένα στρατηγικός πολιτικός διάλογος και κατόπιν τα project, τα έργα. Όμως ε, δεν, υπάρχει δεν υπάρχουν ούτε σύνοδοι κορφής, ε, ούτε διάλογος, ούτε project. Δημιουργήθηκε μια γραμματεία προχωρήσουμε. Όμως η γραμματεία που έχει μικρά project πρέπει να ασχοληθεί και με τον πολιτικό διάλογο διαφορετικά. Δεν ε, έχει νόημα. Για τη δεύτερη ερώτηση του φίλου μου Φίτσας από το όρο που αφορά την ε, Αραβική Άνοιξη. Εγώ νομίζω ότι είναι ουσιαστικά κάτι χωρίς επιστροφή, όχι γιατί δεν υπάρχουν αυταρχικά καθεστώτα, αλλά γιατί οι αραβικές κοινωνίες δεν θα επιστρέψουν στο παρελθόν και θα απαιτήσουν μεγαλύτερη πολιτική, οικονομική συμμετοχή. Και επομένω, αν και δεν δέχονται θεοκρατικές τάσεις ή ριζοσπαστικές ηγεσίε ε, και έχουμε μια διαδικασία αναταραχής, μακροπρόθεσμα, δεν μπορούμε να φανταστούμε κάποιες αραβικές χώρες της Βορειοαφρική που να κυριαρχούνται από αυταρχικά καθεστώντα για πάντα, ακόμα και στην Αίγυπτο με τις δυσκολίε που έχουμε. Ήδη οι πολίτες θέλουν να έχουν την ικανότητα της συμμετοχής, θέλουν να έχουν την αξιοπρέπεια ότι είναι πολίτες και να μπορούν να αποφασίζουν για το μέλλον, για το μέλλον τους. Όμως, προκειμένου να είναι αποτελεσματική αυτή η συμμετοχή και να συνεισφέρει στην ευημερία και τη σταθερότητα των χωρών, θα πρέπει να γίνει με ένα πολιτικό προσανατολισμό, γνωρίζοντας ποιες είναι οι εσωτερικές συνθήκες, ποιες είναι οι δικές τους και οι δικές μας ευθύνες ποιες είναι οι αναγκαιότητές μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά τους. Ε, όπως λέχθηκε το 2011, μας ε, χτυπούν την πόρτα και εμείς έχουμε την δική μας οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν ακούμε. Ήμασταν ε, αφηρημένοι, ασχολούμασταν με άλλα πράγματα. Στα δικά μας, ασχολούμασταν με τα δικά μας θέματα. Γι' αυτό τώρα θα πρέπει να ξαναρχίσει ο διάλογος και ο τρόπος να προσεγγίσουμε την κοινωνία των πολιτών είναι να τη βοηθήσουμε να οικοδομήσει τον δημοκρατικό χώρο και πολιτικό χώρο που χρειάζεται στις κοινωνίες. Τώρα για τον Τραμπ. Η ανάλυση που γίνεται στον αραβικό κόσμο και στην και την ε, Αμερικανική κυβέρνηση είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε για διάφορους λόγους θα δείξουν ε, μια σταδιακή αποδέσμευση από την περιοχή. Υπόθηκε πάντοτε ότι η Μέση Ανατολή και η Αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή ξεκινά από το 1949 με το σύμφωνο της οικογένειας Σαούδ το, με τον πρόεδρο Ρούσβελτ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αποκτούν τον έλεγχο και τον εφοδιασμό του πετρελαίου και του αερίου και οι Ηνωμένε Πολιτείε εγγυώνται την ειρήνη και τη σταθερότητα και έχουμε και τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και την αναγκαιότητα να εγγυθούν και να υπερασπίσουν την ύπαρξη του Ισραήλ. Μάλιστα. Το ενεργειακό θέμα, οι Ηνωμένε Πολιτείε ήδη από την κυβέρνηση του Ομπάμα άρχισαν να δείχνουν την αποδέσμευσή τους. Όλα τα στοιχεία που αναλύθηκαν για τη Συρία, για την ε, μη στρατιωτική παρέμβαση στη Συρία για το ότι δεν σεβάστηκαν οι κόκκινε γραμμέ τους ήδη από την πλευρά του Αμερικανικού establishment ε, ήταν ε, μια βούληση απομάκρυνσης. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπήρχε παρουσία, αλλά όχι η ίδια παρουσία της Αμερικανικής υπερδυναμής. Επομένως ο Τραμπ θα είναι αυτάρκης στην ενέργεια με την υδραυλική ρογμάτωση, δεν θα εξαρτάται από τις χώρες του κόλπου και θα έχει τελικά και ένα δίκαιο με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη και η Ευρώπη θα πρέπει και μπορεί, μπορεί και μπορεί να βρει τον ιστορικό και στρατηγικό της και ηθικό της χώρο. Και πρέπει να προετοιμαστούμε. Θα περιμένουμε τις πρώτες δράσεις της κυβέρνησης Τραμπ που μπορεί να μας λάβουν εξαπίνες. Ίσως ε, μακάρι όχι. Δεν προκρίνω τίποτα, αλλά δεν θα έπρεπε η ευρωπαϊκή διπλωματία να αρχίσει να προετοιμάζεται για κάποιους πολύπλοκους μήνες και δύσκολα χρόνια όπου η αμερικανική παρουσία δεν θα είναι τόσο έντονη, δεν θα αναλαμβάνει την ίδια δέσμευση όπως στο παρελθόν και θα αφήσει να ρέουν τα πράγματα όπως να είναι και να μην επιλύεται τίποτα. Εμείς οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να αναλάβουμε περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο για να περισπίσουμε τα συμφέροντά μας. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν η κυβέρνηση Τραμπ αποφασίσει να μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ την πρεσβεία των ΗΠΑ. Θα περιοριστούμε σε μια δήλωση I'm deeply concerned Λέω μιλητή στα αγγλικά. Ίσως strongly concerned. Very strongly concerned. Ή με κάποιο θετικό τρόπο θα αποφύγουμε να δημιουργηθούν συνθήκες αντιπαράθεσης Όλα αυτά θα πρέπει να δώσουν κίνητρα στην ευρωπαϊκή διπλωματία για να κινητοποιηθεί. Και αυτό με οδηγεί στο να απαντήσω στον κύριο Μαραγάλ, συμφωνώντας απόλυτα με τη θέση του. Η διπλωματία χρειάζεται να έχει ένα μέσο άμυνας και ασφάλειας, αλλά αυτή είναι η εξωτερική πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Εμένα, όταν μιλάμε για διπλωματία, δεν μου αρέσουν τα επίθετα. Μιλάμε τώρα για οικονομική διπλωματία, ψηφιακή διπλωματία, πολιτιστική διπλωματία, δημόσια διπλωματία. Υπάρχει μόνο και μόνο διπλωματία με ένα δέλτα κεφαλαίο, αυτή που ασχολείται με την εξωτερική πολιτική αυτή που ασκεί τη διπλωματία προκειμένου να υπερασπιστεί τα στρατηγικά της συμφέροντα, αυτή που επιλύει σειράξεις και διαπραγματεύεται, που χρειάζεται ένα σκέλος άμυνας και ασφάλειας, αλλά αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι μια διπλωματία επιτόπου Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Τι αιτήματα έχουμε να κάνουμε. Έλεγε ο κ. και είχε δίκιο. Θα θέλαμε να έχουμε μια νέα πολιτική επιτροπή. επιτροπή. και ο ε, ε, κύριος Λέντα και ο κύριος Παπανδρέου και ε, η κυρία Μπενίτα Φεραίρο και ο πρώην Υπουργό τη Μαυριτανία. Όλοι αυτοί οι πρώην Υπουργοί και Πρωθυπουργοί είναι άνθρωποι που είχαν τη σχετική πείρα. Εμείς ευχαρίστως να επανέλθουμε και να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ζητήματα αυτά. Αυτή είναι η άμεση απάντησή μου. Πρέπει να συνεχίσουμε με τη δέσμευσή μας για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, να προσπαθήσουμε να πείσουμε το Ισραήλ ότι είναι απαραίτητη η ειρήνη να δουλέψουμε πάνω σε μια γαλλική πρωτοβουλία, μια οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να επιφέρει σταθερότητα και ειρήνη στην περιφέρεια αυτή. Όλοι μαζί μόνο μπορούμε να κάνουμε κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε Μωρατίνος. Είναι προνόμιο για μας ε, να συζητάμε μαζί σας και να σας ακούμε. Έχουμε καθυστερήσει με τις εργασίες μας. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους διερμηνείς αν μπορούν να μείνουν 10-15 λεπτά ακόμη, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας. Εγώ σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ προς αυτά, Κλέρκ. Πρέπει να μιλήσουμε για τις δικές μας δραστηριότητες. Θα επιστρέψουμε στα δικά μας ζητήματα για λίγο. Ξέρετε ότι στη Ρώμη έγινε η συνεδρίαση του διευρυμένου Προεδρίου που αποφάσισε να συμπληρώσει την ανανέωση των δομών της Επιτροπής μας η Ιταλική Προεδρία συγκεκριμένα αποφάσισε να δώσει προσανατολισμό στις δραστηριότητες των επιτροπών αποφασίστηκε να κάνουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους παρέμβασης, μια σειρά οριζόντιων προτεραιοτήτων για την ε, μετανάστευση και την τρομοκρατία και την ασφάλεια και μια δυνατότητα ότι εμείς σε σχέση με την μεταρρύθμιση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο γρήγορα και γι' αυτό η ομάδα εργασίας υπό την προεδρία της ε, συναδέλφου Μπεκίν παροτρύνεται να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να γίνει μια μεταρρύθμιση τουλάχιστον του οικονομικού κανονισμού έτσι όπως αποφασίστηκε από την Ολομέλεια της Λισαβόνας πριν 1,5 χρόνο σε ό,τι αφορά το σεβασμό των διαδικασιών βρήκαμε μια ρεαλιστική λύση από την πρόταση της Ιταλικής Προεδρίας στην απόφαση του Προεδρείου να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια ε, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο και αποφασίστηκε, είχε αποφασιστεί το πάγωμα στην Ολομέλεια της Λισαβόνας το 2015. Αυτό για ποιο λόγο, γιατί ορισμένες επιτροπές και ορισμένες χώρες βρέθηκαν σε μια κατάσταση αδυναμίας να οργανώσουν τις συνεδριάσεις τους. Οι Τινήσοι δεν είχαν χρήματα για την διερμηνία, για μια συνεδρίαση για το γυναικείο ζήτημα και επίσης και από την πλευρά των Ευρωπαίων υπήρξε αίτημα της Πορτογαλίας να χρησιμοποιηθούν εδώ οι χώροι του Κοινοβουλίου γιατί δεν είχαν τους απαραίτητους πόρους για να οργανώσουν τη συνεδρίασή τους. Η Ιταλική Προεδρία και το Προεδρείο αποφάσισαν επομένως να λάβουν μια πολιτική απόφαση για να ανασταλεί αυτό το μπλοκάρισμα, απόφαση που ελήφθη ομόφωνα από το Προεδρείο. Εμείς υποστηρίξαμε αυτή την ε, πρόταση και μάλιστα είπαμε ότι όπου είναι απαραίτητο θα δώσουμε μια νομική βοήθεια από το Γραφείο του Κοινοβουλίου προκειμένου να ξεκαθαριστούν ε, διάφορα προβλήματα που είναι από την βάση της Λισαβόνας. Θα έλεγα ότι αυτά είχα να σας πω. Αν ε, κυρία Μπικίν θέλει να προσθέσει κάτι, έχει το λόγο. Και κατόπιν όποιος άλλος θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε σας όλοι για τόσο είπατε. Εμείς προσπαθούμε να προχωρήσουμε ως ομάδα εργασίας για τη μεταρρύθμιση της ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης και φυσικά για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό θα έπρεπε να προχωρήσει παράλληλα. Υπάρχουν όμως κάποιες δυσκολίες γιατί όλες οι συνεδριάσεις ε, ουσιαστικά είχαν ελλειπή συμμετοχή και μάλιστα και στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου ε, εκπροσωπούνταν τέσσερις από τις πέντε επιτροπές αλλά μόνο ε, λίγα μέλη. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσαμε να έχουμε επικοδομητική συζήτηση. Γι' αυτό το λόγο στείλαμε και ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να έχουμε πιο ρεαλιστικές εργασίες με μία ημερομηνία λήξης ε, ως τις 15 ε, Νοεμβρίου. Δεν έγινε σεβαστή βέβαια αυτή η προθεσμία παρά από τη Γαλλία, την Πορτογαλία. Η κυρία Ροντρίγες μας το έστειλε, την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και βέβαια αυτό δεν αρκεί για να προχωρήσουμε για αυτόν τον προβληματισμό. Επομένω, θα ξανακάνουμε αυτή τη διαβούλευση και θα σα τηρούμε ενήμερου για το αποτέλεσμα. Σίγουρα θα έχουμε και με επόμενη συνεδρίαση το Γενάρη. Και θα ήθελα και να με βοηθήσετε όλοι για να μπορέσουμε να έχουμε μια καρποφόρο συνεδρίαση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα της συνεδρίσης του Προεδρείου, πρόκειται για ένα διευρυμένο Προεδρείο στις 22 Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της διαδικασίας έχουν αρθεί οι δικές μου τα δικά μου ερωτηματικά. Δεν ε, μπορεί ουσιαστικά να ανατραπεί μια απόφαση που έχει ληφθεί από την Ολομέλεια. Τώρα, στην περίπτωση αυτή για την πολιτική απόφαση, εγώ μπορεί να συμφωνώ, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι μια προσέγγιση που μπορεί να ζημιώσει τη συνέχεια των εργασιών μας. Γιατί ακριβώς πρόκειται για θέματα τα οποία δεν ξέρουμε στη συνέχεια πώς μπορεί να ερμηνευτούν από τους όλους συναδέλφους. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό αυτό, όπως προτάθηκε και από τον κύριο Σεσόλη στη Ρώμη, να θέσουμε το ζήτημα στην νομική μας υπηρεσία και στη συνέχεια σε όλα τα κοινοβούλια μέσω της γραπτής διαδικασίας. Είναι ένα σύστημα ε, ένα σύστημα με εκπαιδευτικές προεδρίες ε, ουσιαστικά ε, καθιστά επικίνδυνο στο να αναιρέσει ένα προεδρείο απόφαση μιας ολομέλειας. Θα μπορούσε αυτό να βλάψει λοιπόν την συνέχεια των εργασιών μας και να προκαλέσει δυσκολίες. Όμως νομίζω ότι αν έχουμε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε και με γραπτή διαδικασία. Σημειώνω λοιπόν την απόφαση της Ιταλικής Προεδρίας και σε ό,τι αφορά τις εργασίες θα προσπαθήσαμε εμείς να είμαστε όσο πιο επικοδομητικοί και φυσικά όλες οι αποφάσεις και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και του νέου δημοσιονομικού κονισμού θα πρέπει να συζητηθούν στην Ολομέλεια. Θα συζητηθούν ε, ίσως ε, στην επόμενη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου στο Προεδρείο, όμως ε, και πάλι η απόφαση θα ληφθεί το Μάιο. Μάλιστα, επόμενος ομιλητής. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο, όχι. Απλά για να προσθέσω κάτι. Σας ευχαριστώ κύριε Μπινίν για τα όσα είπατε. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρό οι βουλευτές ε, που έχουν δεσμευτεί να συμμετέχουν σε μια ομάδα εργασία να μην συμμετέχουν ποτέ. Είναι λάθος κάτι τέτοιο. Δεν λειτουργούν ε, τα διάφορα όργανά μας και στην Λισαβόνα είχαμε ε, πει ότι θα Είχαμε αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και κατόπιν στην πορεία μιλήσαμε και για μεταρρύθμιση ολόκληρη τη κοινοβουλευτική συνέλευση τη Μεσογείου. Και αυτό το έργο που το ανέλαβε η Επιτροπή της κυρίας Μπεκίν δεν μπορεί να υλοποιηθεί επειδή δεν συμμετέχουν οι βουλευτές. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πιστεύω ότι η Προεδρία θα πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σχετικά με το θέμα προκειμένου να επιτρέψει στην ε, συνέλευση της Μεσογείου να σεβαστεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει. Και από τη δική μου σκοπιά, αν ε, δεν υπάρχουν αντεμβήξεις, εγώ πιστεύω ότι η Προεδρία θα πρέπει να παρεμβαίνει με ένα κάθετο τρόπο. Σε ό,τι αφορά την ε, απόφαση να υπερβληθεί αυτό το μπλοκάρισμα, γιατί ουσιαστικά συνέβη επειδή υπήρχαν κάποιες υλικέ δυσκολίες, σας ανέφερα την περίπτωση των Τινσίων και των Πορτογάλων που είχαν κάνει κάποια αιτήματα, θα πρέπει ουσιαστικά οι επιτροπές να είναι σε θέση να λειτουργούν και γι' αυτό ελήφθη μια απόφαση και φυσικά αν υπάρχουν παρατηρήσεις θα τις υποβάλουμε και στη νομική μας υπηρεσία προς έγκριση όμως ε, αυτά εντός μηχανισμών που ρυθμίζουν την χρήση των πόρων αυτών. Και <laughs> είναι κάτι πολύ απαιτητικό. Εδώ μιλάμε για επιπλοκή 90.000, αποδέσμευση 90.000 ευρώ που θα επιτρέψουν στους τινήσιους να πληρώσουν τη διερμηνία ή στους Πορτογάλους να νοικιάσουν ε, ένα χώρο για τη συνειδρίαση. Κύριος Φίσας, Πρόεδρε, καθώς ε, ε, μιλάμε για τη συμμετοχή, νομίζω ότι εσείς ο αρμόδιος να το θέσεις αυτό. Μερικέ φορέ υπάρχει πρόβλημα όταν έχουμε την πράσινη εβδομάδα και υπάρχει, παραδείγματο χάρη, ένα ταξίδι τη Γερομέντη ή κάποια άλλη αντιπροσωπεία και συμπίπτει με συνεδρίαση άλλων επιτροπών, με την ΙΝΤΑ, παραδείγματο χάρη κτλ. Γιατί εγώ τι κάνω, είμαι σε δύο επιτροπέ και δεν γίνεται την ίδια εβδομάδα να είμαι σε δύο μέρη. Αυτό είναι πρόβλημα λοιπόν. Και δεν ξέρω πώ μπορούμε να το λύσουμε. Πρόεδρο, εγώ πιστεύω ότι αυτό Μπορούμε να το λύσουμε μέσω της δομής μας καταρχήν και με τη δυνατότητα να έχουμε μία οργάνωση και τα χρονική στιγμή που να λαμβάνει υπόψη τα ταυτόχρονα καθήκοντα των βουλευτών. Ίσως να βρούμε έναν τρόπο για να διαχειριστούμε αυτές τις δυσκολίες. Εγώ πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να συμμετέχουμε. Αλλά βέβαια εσείς είστε αυτοί που συμμετέχετε πάντα στις συνεδριάσεις ε, της συνέλευσης. Θα πρέπει ουσιαστικά να είμαστε κάποιες προαυστηροί απέναντι σε αυτούς που δεν συμμετέχουν, ε, γιατί τελικά μπλοκάρεται η δραστηριότητά μας. Ακόμα ακούσαμε σήμερα τον κύριο Μωρατίνος και ναι, ναι. αν δεν έχουμε στη συνέχεια δυνατότητα να διατηρήσουμε ζωντανή αυτή τη φλόγα του διαλόγου, νομίζω ότι τελικά όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη αξία. Στην ε, Λισαβόνα πιθανότητα αξιολογήθηκε αυτό το θέμα και νομίζω ορθά ότι ήταν ε, το θέμα του να ληφθεί με απόφαση για τον προϋπολογισμό για να υπάρχει μια μεταρρύθμιση, όχι για την εμπλοκή. Στην πραγματικότητα, αυτό τον 1,5 χρόνο εμείς δεν δώσαμε συνέχεια σε εκείνη την απόφαση. Και πιθανότατα, λόγω όσων είπε η κυρία Μπεγκίν, επειδή δεν υπάρχει υπαρκή συμμετοχή των βουλευτών στην ομάδα εργασίας που πρέπει να παρουσιάσει αυτή η μεταρρύθμιση. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πιστεύω ότι η Προεδρία και ο Πρόεδρος Σούλτς ε, θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις. Ε, noi, ε, per quanto riguarda mm, poi eh, giudizio... Σε ό,τι αφορά τώρα την κρίση που έγινε στη Ρώμη, την απόφαση που ελήφθη, εγώ νομίζω ότι στη μεταρρύθμιση στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση των ε, κλιματοοικονομικών μηχανισμών θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε συνεισφορά από τις χώρες. Δεν μπορούμε όλα να τα φορτώσουμε στις προεδρίες ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Αν κάτι είχαμε αποκτήσει από την συνέλευση της Μεσογείου και ιδίω από την Πορτογαλική Προεδρία, μάλλον από την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήταν ε, αυτό να ευνοηθεί η οικονομική συμμετοχή όλων των χωρών. Όμω αυτό θα πρέπει να το κάνουμε εμεί σε ένα ισχυρό σημείο, όχι σημείο αδυναμία. Ελήφθη η απόφαση στη Λισαβόνα, όμω εμεί πρέπει να αναπτύσσουμε και τι δικέ μα πρωτοβουλίε και όλε οι χώρες ε, να μπορούν να υλοποιούν τι συνεδριάσει του και τι συνεδριάσει των επιτροπών. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα το ορθό. εμείς στην επόμενη συνεδρίαση. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με την υπατή εκπρόσωπο. Αυτό είναι ραντεβού το οποίο όλοι το περιμένουμε, μια συνάντηση που όλοι το περιμένουμε, γιατί έχουμε ζητήματα που ξανανοίγουν στη Μεσόγειο. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που μας αφαιρούν. Στο Στρασβούργο, το επόμενο Φεβρουάριο θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση. Είναι το μεταξύ, ελπίζω ότι οι επιτροπέ και ομάδε εργασία θα μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Σα ευχαριστώ.